Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε τις εργασίες της Συνόδου και θα αρχίσω να μιλάω στα Ουγγρικά. Το πρώτο θέμα απόψε Λοιπόν, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Μπέντσεν, σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Θα δώσω αμέσως το, ρόλο, το λόγο στον εισηγητή, κύριο Μπέντσεν, που θα λάβει το λόγο για δύο λεπτά. Thank Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή απόδοση το 2020 και το σχέδιο δράσης της Ένωσης δείχνει ότι και 10-11% να φτάσουμε θα είναι αρκετά καλό γιατί θα μπορέσουμε να... να οδηγήσουμε την ενεργειακή απόδοση για πολλούς λόγους. Και βεβαίως ο στόχος αυτός απαιτεί να χρησιμοποιήσουμε μικρότερη ενέργεια. Άρα υπάρχει εξοικονόμηση τις ε, ενέργειες για την επίτευξη του στόχου του 20% μέχρι το 2020. Η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Εμείς ωστόσο είμαστε πιο καθυστερημένοι. Παρακολουθούμε την Κίνα και άλλα κράτη που επιδότησαν την βιομηχανία στις Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχουν σοβαρά κονδύλια για αυτό ενώ στην Ένωση σκενόμαστε μόνο την ε, εξοικονόμηση και όχι την απόδοση. Σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να σταθούμε σε ορισμένους στολείς που ενώ ξεχνάμε ότι πρέπει να ε, έχουμε αποτελέσματα οικονομικά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά μας. Η ενεργειακή απόδοση φέρνει και θέσεις εργασίας, δουλειά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό είναι πολιτική ε, πλάνο δράσης, πολιτικές ε, εξοικονόμησης και, και κίνητρα. Είναι διαφορετικές δραστηριότητε. Τα εθνικά προγράμματα δεν έδειξαν ότι είναι εξαιρετικά αποδοτικά, έχουν όμως ε, μεγάλες δυνατότητες. Είναι αναγκαίο λοιπόν να μπορέσει η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα καταλληλότερα εργαλεία και να απορρίψει, να απορρίπτει προγράμματα δράση αν δεν είναι πολύ φιλόδοξα. Κάτι που σημαίνει και διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία των χωρών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποφασίσουν χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις τους. Σε κάποιες χώρες η δυνατότητα ενεργειακής εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες. Άλλες χώρες θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε εξοικονόμηση στην παραγωγή ή στη βιομηχανία. Κατόπιν υπάρχουν ε, πρότυπα και σήματα. Τα πρότυπα είναι πολύ σημαντικά διότι δείχνουν την δυνατότητα εξοικονόμησης και την ανάγκη βελτίωσης των και καινοτομίας. Τώρα, η στεγαστική πολιτική είναι πολύ σημαντική επίσης ένα μεγάλο το τμήμα της κατανάλωσης προέρχεται από τα κτίρια, ε, τομέα όπου μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ε, εξοικονομήσεις. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι τομείς αυτοί θα μπορέσουν να συμβάλλουν για μια καλύτερη ανταγωνιστικότητα και τα επόμενα έτη. Συστήνουμε λοιπόν να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπου οι επενδύσεις επαναλαμβάνονται συχνά μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο την δραστηριότητα αυτή και ελπίζω η έκθεση να εκκληθεί ε, με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη και για την, ε, τις επιχειρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Ότιγκερ. Παρακαλώ, εξ ονόματος της Επιτροπής. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τρεις αυτές επιτροπές ε, δούλεψαν ε, πολύ αποδοτικά και είμαι ιδιαίτερη ευγνώμων πως αυτές ιδιαιτέρως ε, προς τον κύριο Μπέντσεν αλλά και προς άλλους βουλευτές που έχουν ασχοληθεί για πολύ καιρό με το θέμα αυτό. Ε, ο στόχος του 23% 23% του 23% όσον αφορά την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση της ενέργειας μελλοντικά. Ε, βρίσκονται, υποδεικνύουν το σωστό δρόμο. Και αν ε, δεν ε, διαπραγματευτούμε θα αστοχήσουμε. Δηλαδή έχουμε κάποια πρότυπα, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, το... και η Κομισιόν, αλλά οι εξελίξεις μετά την κρίση δεν ε, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση του 20% αλλά το πολύ 8 ή 9% για τα προσεχή χρόνια. Αυτό είναι ένας εφικτός στόχος. Τώρα, όσον αφορά την έννοια ενεργειακή αποδοτικότητα, δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχη, γιατί δεν μπορεί να την καταλάβει κανεί εκτό από εμά. Εάν ρωτήσετε τους γειτονέ σας ή τους φίλους σας τι σημαίνει αυτή η έννοια. Η έννοια τη εξοικονόμηση ενέργεια είναι ε, γνωστή, αλλά όχι έννοια της ενεργειακής αποδοτικότητα. Και πράγματι όσον αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου, ε, το ερώτημα τι θα πρέπει να επιτευχθεί εδώ δεν είναι παρκώς ε, ορισμένο. Έχουμε ένα απολογισμό όσον αφορά την ενέργεια και ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό κατανάλωσης της ενέργειας εάν δούμε τα πράγματα από μια εξέλιξη της κατανάλωσης της ενέργειας βλέπουμε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ανωδική και χωρίς ε, ενεργειακή αποδοτικότητα θα συνεχίσουμε να έχουμε μία αύξηση στην ε, κατανάλωση της ενέργειας. Στη Γερμανία όχι αλλά σε άλλες χώρες ναι, λόγω των ε, ηλεκτρικών ε, κινητήρων, της ε, βιομηχανικής ανάπτυξης εν γέννη κλπ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανείς καμία αντικειμενικά ισχύουσα προοπτική. Δηλαδή το 20% ποιας ποσότητας ενέργειας. Αυτό είναι άγνωστο. Ποια θα είναι η κατανάλωση ενέργειας. Και εγώ θεωρώ ότι οι προγνώσεις και οι αριθμοί εδώ είναι αμφισβητούμενοι. Γιατί ορισμένοι λένε ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχει μια ξεκάθαρη ανωδική ε, τάση όσον αφορά την ε, δαπάνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοιχεία, αξιόπιστου αριθμού. Θέλουμε μέχρι το Φεβρουάριο και Μάρτιο να επεξεργαστούμε αυτά τα αξιόπιστα στοιχεία. Οι επικεφαλεί των κυβερνήσεων το Φεβρουάριο θα πρέπει να πάρουν εξίσου σοβαρά το θέμα όπως και πριν από την κρίση. Γιατί έχω την άποψη ότι η κατάσταση των πραγμάτων σήμερα όσον αφορά του δεσμευτικού στόχου για τι χώρε μέλη ε, δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένα τα μέλη να υπερψηφίσουν αυτούς τους στόχους. Ε, Εμείς είμαστε, ε, γιατί βρισκόμαστε ακόμα σε μεγάλη απόσταση από τη δεσμευτικότητα των στόχων που είχαν αποφασιστεί πριν από δύο ή τρία χρόνια. Δηλαδή, ποια είναι η συνυπρογνώση του 2020 χωρίς ενεργειακή αποδοτικότητα. Μία θεωρητική θεώρηση και στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται με το μείον 20%. Λοιπόν, το θέμα είναι πού βρισκόμαστε. Καταρχήν όσον αφορά τα κτηριακά αποθέματα, όσον αφορά την κατοικία, την εργασία και τη βιομηχανία. Εδώ ε, στα κτίρια πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και εδώ θα πρέπει να εργαστούν οι δήμοι, οι κοινότητες, ε, τα κρατήδια εδώ όπου το δημόσιο έχει μία κυριότητα θα πρέπει η αποδοτικότητα να είναι πρώτη στο στόχος. Δεύτερον, έχουμε τα διαφορετικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εδώ στις διάφορες χώρες υπάρχουν διαφορετικά μεταξύ τους ε, προγράμματα εξυγίανσης τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν και να συντονιστούν θα πρέπει ίσως να χρηματοδούμε λιγότερα λιθόστρωτα για δημόσιες πλατείες και λιγότερες παρκαμπτήριους οδούς και ε, ε, να συγχρηματοδοτήσουμε περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί αυτός είναι ένας καθοριστικός στόχος και για, τον επόμενο, για την επόμενη περίοδο προϋπολογισμού για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα το θέμα μεταφορές. Ε, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη όπου για χίλιους ε, ε, κατοίκους αντιστοιχούν 550 ιδιωτικά οχήματα ενώ σε άλλες χώρες μόνο 120. Θα υπάρξει μια εναρμόνιση, αλλά όχι 100 για οχήματα για χίλιους ε, κατοίκους. Όχι, χρειαζόμαστε περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα για τις μεταφορές. Η μεταφορά η οποία ε, αποφεύγεται είναι η πιο αποτελεσματική εδώ. Αυτή η αρχή ισχύει. Τώρα, όσον αφορά την ε, βιομηχανία. Ε, εδώ υπάρχει το θέμα της δημοσιογότητας των στόχων ε, προτεραιότητα. Στο Συμβούλιο Ενέργειας, ε, σε ένα άτυπο γεύμα, θέσαμε το σχετικό ερώτημα. Και θα πρέπει να σας πω ότι οι χώρες μέλη και οι Υπουργοί Ενέργειας, όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, είναι αρκετά ευαίσθητοι και δεσμευμένοι, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμοι για τη λήψη αποφάσεων σε σχετικά με δεσμευτικούς στόχους. Σκεφτείτε ένα μια χώρα μέλος όπως η Πολωνία. Μείον 20% θέτω το ερώτημα. Ή μια, ένα κορισμένο μέλος όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία. Πώς θα τα καταφέρουμε, για παράδειγμα, η Αυστρία και η Γερμανία δέχονται το μείον 20% ούτως ώστε η Πολωνία να μπορεί να χρηματοδοτήσει τη δική της ε, ανάπτυξη και να προσαρμοστεί όμως ε, στους στόχους αυτούς. Εδώ ε, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές συζητήσεις ως φορά συγκεκριμενοποίηση σε όπως είναι η μεταφορά, η κατοικία, ε, και στο επίπεδο των διαφόρων χωρών μελών. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και θα ήθελα στις 4 Φεβρουαρίου να απασχολήσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το θέμα αυτό, ούτω ώστε να δούμε πολύ συγκεκριμένα πόσο σοβαρά προτίθενται οι κυβερνήσεις να πάρουν αυτό το στόχο και θα θέλαμε να υποβάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο για μια νέα, ένα νέο σχεδιασμό ενεργειακής αποδοτικότητας και να σας τον υποβάλουμε. Και ασφαλώς την Άνοιξη και το καλοκαίρι θα έχουμε παρκώς την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και η δεσμευτικότητα των στόχων. Γιατί ενδεχομένως ε, το μέτρο της επικουρικότητας ε, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ένα σχέδιο δύο βαθμίδων. Ε, η πρώτη βαθμίδα ε, σε εκούσια, δηλαδή σε εθνικό επίπεδο ετήσια σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητας. Και λέμε τι περιαναμένουμε έτος ανά έτος. Αλλά δεν αναμένουμε την επίθεση του στόχου μείον 20% μετά από δύο χρόνια αλλά αναμένουμε μια δεσμευτικότητα εάν δούμε ότι τα πρώτα δύο χρόνια στην φάση της εκούσιας δέσμευσης δεν έχουμε απτά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Τώρα ξεκινούμε με τις παρεμβάσεις εξ ονόματος των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο κύριος Λίσε πρώτος για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, μας κυρίε και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια διάθεση στη γερμανική μετάφραση ε, που λέει ότι είμαι ο πρόεδρο τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. Δεν ισχύει, είμαι ο εισηγητή. Αλλά υπό την έννοια αυτή θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπέντσεν για την πολύ καλή εργασία που έκανε και για την καλή συνεργασία με εμά. Πραγματικά διατύπωσε μια φιλόδοξη στρατηγική όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το πιο ε, φτηνό μέσο για να μειωθούν οι σπατάλε ε, σε, ενέργεια και να μειωθούν οι εισαγωγές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να στερφόμαστε προς την Ρωσία ή άλλες ε, χώρες. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος συνέταξε μια περιεκτική έκθεση μια... όπου ε, δεν θα ήθελα να επαναλάβω όλους τους φιλόδοξους στόχους, αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, και μιλήσαμε σχετικά κύριε Επίτροπε, ε, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει ε, μακρόπνοους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Γιατί αν κάνουμε ένα σχεδιασμό για το 2050 θα πρέπει να ξέρουμε πώς καταναλώνουμε περίπου. Και δεύτερον, όσον αφορά τον ορισμό. Επισημάναμε τις σχετικές δυσκολίες και θεωρώ ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς, το, προς την ποσότητα της κατανάλωσης της ενέργειας. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεν έχουμε ε, στοιχεία κατά τα άλλα. Και ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά στη στρατηγική που θα διαβάσουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ για την ε, Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Η κυρία Κολάζ Καμπομπίσκα έχει το λόγο 1,5 λεπτό και αυτή. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή απόδοση είναι μεγάλη πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσει τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αποτελέσει ε, στοιχείο κλειδί της στρατηγικής μας αυτό το σχέδιο δράσης. Σήμερα ετοιμάζουμε ωραίες εκθέσεις και λέμε ότι τα κράτη-μέλη αν προωθούν και εφαρμόζουν την πολιτική που έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όμως αντιλαμβανόμαστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα δεν είναι δυνατόν να μετρήσουμε επακριβώς τις προόδους που έχουν σημειωθεί. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να καθορίσουμε συγκεκριμένους στόχους αν βασιστούμε στα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή που δεν είναι επαρκώς ακριβή. Χρειάζονται λοιπόν νέες τεχνολογίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας. Και πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Στην Κοπενχάγη η κατάσταση δεν είναι ίδια με αυτή που ισχύει στην Ανατολική Πολωνία. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε παντού τα ίδια σχέδια δράσης. Χρειαζόμαστε σχέδια δράσης που να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει και αυτή να λάβει μέρος σε όλη αυτή την προσπάθεια. Χρειάζεται συντονισμός σε ε, επίπεδο κράτους μέλους με τις αυτοδιοικητικές αρχές διότι αλλιώς οι προσπάθειες δεν θα αποδώσουν και θα, το όλο, θα στεφθεί με αποτυχία το όλο εγχείρημα. Ευχαριστώ. Προχωρούμε στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Ρόιλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνου οι οποίοι δούλεψαν πάνω σε αυτή την έκθεση, ιδιαίτερα τον συνάδελφο κ. Μπέντσεν. Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία τη έκθεση, και ίσω να κάνω κάποιου προβληματισμού εδώ. Συμφωνούμε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα, η, η ενεργειακή εξοικονόμηση δεν μπορεί παρά να είναι η λύση, η πιο απλή και η πιο λογική. Το θέμα είναι πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο. Και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα τι μας απέφερε εδώ στο Κοινοβούλιο το να θέτουμε όλο και υψηλότερα ποσοστά. Ε, καταφέραμε περισσότερα πράγματα, μπορέσαμε να κινήσουμε περισσότερα πράγματα. Ή, πού έγινε ακριβώς αυτή η οικονομία της ενέργειας. Γιατί μου λένε ότι η βιομηχανία η οποία καταναλώνει πολλή ενέργεια ε, εξοικονομεί ε, περισσότερη ενέργεια γιατί αυτό τη συμφέρει περισσότερο αλλά ε, τι γίνεται με τους πολίτες όταν γνωρίζουν ότι μια συσκευή ε, χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, ίσως δεν θα τη χρησιμοποιήσουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η μέθοδος να δουλεύουμε ποσοστά, αλλά να παρέχουμε κίνητρα. Δεύτερον, ο κύριος Επίτροπος είπε πολύ ξεκάθαρα πόσο πολύπλοκη είναι και μόνο η περιγραφή αυτή τη έννοια. Περί τίνο πρόκειται και πώ διαμορφώνονται τι διάφορε χώρε μέλη. Η συνάδελφο είπε ότι οι χώρε μέλη έχουν εντελώ ε, διαφορετικά συστήματα. Ε, είναι σωστό να ορίζουμε ένα δεσμευτικό ποσοστό ή θα πρέπει να κάνουν περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι σε επίπεδο τη πολιτική θα πρέπει να αποδεσμευθούμε από τι συζητήσει του παρελθόντο που ακριβώ δουλεύουν πάνω σε δεσμευτικού ε, αριθμού και θεωρούν ότι μπορούν ε, να βρουν κάποιε συνταγέ. σω θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο πιο διαφοροποιημένων απαντήσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ε, διαφορές μεταξύ των χωρών και τις αποχρώσεις. Γιατί το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα και όχι ε, η δική μας ε, βολή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόμποντ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Έχω ένα ερώτημα προς τον Σανάλφα κύριο Ρόιλ. Δεν είναι δυνατόν σε μια εξέλιξη να τεθούν δεσμευτικοί αλλά διαφοροποιημένοι στόχοι, γιατί αντιπαραθέσατε ε, δεσμευτικό και διαφοροποιημένο. Νομίζω ότι είναι δύο όροι συμβατοί. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει με κάποια βήματα που προσθέσει ο κ. Επίτροπο. σω μπορούμε να βρούμε έναν δρόμο που κανεί κάνει τι διαφοροποίησει ανά γεωγραφική θέση κάθε χώρα κλπ. Και, από την άλλη μπορεί να ορίσει δεσμευτικού στόχου. Σα ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Συγγνώμη. Κύριε Ρόιλ, θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Και εγώ είμαι υπέρ των διαφοροποιημένων λύσεων και σκέφτομαι πώς θα τα καταφέρουμε να έχουμε αυτές τις διαφοροποιημένες λύσεις. Δεν θα πρέπει να αποκλείουμε ε, το τι πρέπει να κάνουμε πώς. Αλλά σήμερα θεωρώ ότι είναι εσφαλμένο να θέτει κανείς ε, δεσμευτικά νούμερα αριθμούς. Εγώ θα ήθελα να προβληματιστούμε περισσότερο για το πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι βήμα προς βήμα. Και λυπούμε που δεν καταφέραμε περισσότερα πράγματα. Ίσως γι' αυτό θα έπρεπε να επιλέξουμε ένα άλλο δρόμο. Ευχαριστώ. Όπως έλεγα προηγουμένω για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες έχει το λόγο για δύο λεπτά η κυρία Τόμσεν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ξεκινώ ευχαριστώντας ε, τον κύριο Μπένσεν και τους άλλους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή. Πετύχαμε μια συμφωνία σε πολλά θέματα και πετύχαμε ένα στόχο μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Υπήρξαν βέβαια και κάποιες διαφωνίες σε ό,τι αφορά τις τα δεσμευτικά νούμερα. Εμείς συμφωνούμε πρέπει να καθορίσουμε τουλάχιστον έναν στόχο αξικονόμησης 20% καλύτερης απόδοσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη, ε, οικονομία, βιώσιμη που θα δώσει ένα εκατομμύριο νέε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο στόχο αυτός να είναι δεσμευτικό στα κράτη-μέλη. Γιατί βλέπει ότι, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει επιμονή μου βάσεω στόχου που δεν υλοποιούνται ποτέ ακριβώ γιατί δεν είναι δεσμευτικοί. Αντίθετα, όταν θέτει δεσμευτικού στόχου, αυτοί υλοποιούνται. Αυτό ισχύει και φαντάζομαι θα ισχύσει και για την καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Προφανώ με άλλους, συνοδεύοντας την με άλλους στόχους, ε, ε, μικρότερο κόστος για τον χρήστη κυρίω. Σε ό,τι αφορά το κόστος, αυτό θα ήταν πλεονέκτημα για πάρα πολλού πολίτε που υποφέρουν από την ενεργειακή παινία, η οποία πλήττει άτομα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν μεγάλο τμήμα του εισοδήματός τους για τη θέρμανση των οικειών. Δεν υπάρχει ωστόσο κοινό ορισμός για την ενεργειακή παινία και άρα δεν υπάρχουν προσπάθειες για τη μείωσή της. Ε, οι συνέπειες αυτής της παινίας είναι καθοριστικές για την υγεία και για την, και τις συνθήκες ζωής των χαμηλών εισοδημάτων. Εμείς λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση ε, χρηματοδοτώντας ε, την ενεργειακή απόδοση για τις απευθείας της οικογένειας. Με ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης. Ευχαριστώ. Και να ενισχυθεί βεβαίως η μάχη κατά της, ε, υπέρ της ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ. Για την ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών, η κυρία Χολ. Δύο λεπτά. Πρόεδρε, Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Πένσεν, ο οποίο εργάστηκε σκληρά για αυτή την έκθεση. Συνεργάστηκε με τις, συνεργαζόμενος με τους σκιώδεις αιγητές, ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο με το οποίο όλοι συμφωνούν και γι' αυτό το συγχαίρουμε. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση. Η κλιματική ε, αλλαγή μας έχει δείξει ε, ότι η ενέργεια είναι ο καλύτερος, η πρώτη, ο πρώτος τομέας ο οποίος θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τον στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Αλλά δυστυχώς εξακολουθούμε ακόμα να χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Τώρα που είναι ε, αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας η ενέργεια, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πρακτικά προβλήματα που ε, βρίσκουν μπροστά τους οι άνθρωποι προσπαθώντας να, να παραμείνουν σε ένα ζεστό περιβάλλον σε κτίρια και σε οικίες που δεν έχουν την επαρκή μόνωση και αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης. Λόγω λοιπόν αυτής της κατάστασης το 20%, ο στόχος του 20% ενεργειακής απόδοσης είναι μέρος του πακέτου 2020 που φαίνεται ότι οδηγείται προς την αποτυχία, όπως είπε ο Επίτροπος. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 9% ως στόχο θα πετύχουμε σε σχέση με το 20% που έχει προβλεφθεί για το 2020. Έφτασε λοιπόν η στιγμή να παραδεχθούμε ότι κάναμε λάθος το 2008 και πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και να βρούμε πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Μας είπε τι προετοιμάζει για την επόμενη χρονιά ο Επίτροπος και έφτασε η στιγμή να ληφθεί πλέον μια πολιτική απόφαση. Χρειαζόμαστε δεσμευτικό στόχο για την εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλιώς υπονομεύουμε κάθε τι που κάνουμε για την οικονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κύριε Χολ, ο κύριος Ζαντό για τους πράσινους έχει το λόγο με τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Φυσικά θα συγχαρώ πρώτα τον εισηγητή για την ποιότητα της δουλειάς του και θα υποστηρίξω την έγκριση της ε, έκθεση όπως ε, ε, ε, ψηφίστηκε στην Επιτροπή ΤΡΕ αύριο. Υπάρχουν τεράστιε δυνατότητε που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργεια. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λέει αυτό. Αν καταφέρουμε να περιορίσουμε κατά 20% την σπατάλη ενέργεια θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εκατομμύρια θέσεις απασχόληση. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε σε κάθε ευρωπαϊκό νοικοκυριό 1000 ευρώ και να περιορίσουμε βεβαίω τον εξωτερικό ενεργειακό μα λογαριασμό. 20% απόδοση ή μείωση κατανάλωση ενέργεια στην Ευρώπη σημαίνει 15 ναμπούκο, 20% 15 ναμπούκο στον ενεργειακό τομέα και δυστυχώς δεν θα πετύχουμε το στόχο μας, όπως το είπε και η Φιώνα Χολ θέλω, είμαι έτοιμος να μου πείτε ότι δεν κάνουμε σωστά υπολογισμούς και ότι υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες λένε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας το 2020. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει. Η, προ, προσέγγιση για το co-design και το co-labeling των οχημάτων, eco-design και co labeling των οχημάτων δεν φαίνεται να φέρνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε, όταν μας λέτε ότι ότι έχουμε πρόβλημα για τον ορισμό της ενεργειακής απόδοσης, ίσως από θεωρητική άποψη να ισχύει αυτά, αλλά το κλίμα ενέργεια πακέτο είναι πάρα πολύ σαφές ως προς το στόχο. 20% της κατανάλωσης ενέργειας μείωση σε σχέση με τη μια γραμμή βάσης. Δεν είναι θέμα ορισμού της ενεργειακής απόδοσης. Υπάρχουν αυτό που πρέπει να ξεπακέτο, κλίμα, ενέργεια. Μας λένε ότι δεν χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι αυτό ισχύει για, τους, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από λίγες μέρες διαπραγματευόταν στην Κανκούν μια δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, προσπαθώντας να υποστηρίξει το πρωτόκολλο του Κιώτο και εδώ επαναλαμβάνουμε τα επιχειρήματα της Κίνας των ΗΠΑ λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει τίποτα δεσμευτικό. Και αν αντιληφθούμε κάποια μέρα ότι δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας, τότε θα εφαρμόσουμε δεσμευτικά μέτρα. Σχετικά με την έκθεση, ορισμένοι βουλευτές πρότεινα να ενισχυθεί το θέμα της απόδοσης των κτηρίων διότι αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να αναλάβουμε σημαντικέ πρωτοβουλίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με, την, με την ε, βελτίωση και την καλύτερη μόνωση των κτηρίων μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι 40%. Το, οι πολίτες πληρώνουν ακριβά την ενέργεια που καταναλώνουν και αν η ενέργεια είναι πιο ακριβή σε διεθνές επίπεδο θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο Σας παρακαλώ λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να επιμείνετε στον κύριο Βαν Ρομπέου ώστε το ραντεβού της 4η Φεβρουαρίου να είναι και ένα ραντεβού για την κατανάλωση ενέργειας. Ο ειδικό χάρτης που προτείνεται σήμερα από την άποψη αυτή είναι παντελώ ανεπαρκής. Ε, ευχαριστώ πολύ. για τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κ. Σιμάνσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ τον εισηγητή που δούλεψε με ανοιχτό και επικοδομητικό τρόπο για την προετοιμασία της έκθεσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Η ύπαρξη δεσμευτικών στόχων στην ενεργειακή απόδοση είναι κάτι απαράδεκτο για τη δική μας ομάδα. Δεν υπάρχει κοινή μεθοδολογία για τη μέτρηση της πρόοδου που επιτυγχάνεται, ούτε οι δείκτες είναι οι ίδιοι. Πιστεύω ότι η πρόοδος που επιτυγχάνεται θα πρέπει να κρίνεται από τα ίδια τα κράτη-μέλη, διότι ε, η εξοικονόμηση ενέργειας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, πετύχαμε να βελτιώσουμε κατά 10% την απόδοσή μας το 2010. Ωστόσο, βρισκόμαστε στον μέσο ευρωπαϊκό όρο παρά τα αυτά, η Πολωνία δηλαδή. Ένας ενιαίος δεσμευτικός στόχος για όλους θα ήταν καταστροφικός και θα δημιουργούσε ανισάντητες. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Για την Γκουέ το λόγο έχει τώρα η κυρία Ματίας. Δύο λεπτά, δυόμιση λεπτά συγγνώμη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνώ και εγώ ότι η στιγμή που υποβάλλεται η πρώτη αναθεώρηση του προγράμματο δράση για την ενεργειακή απόδοση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Πιστεύω ότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα δεν θα είχε φτάσει να γίνεται αν είχαμε λάβει αυτό νωρίτερα υπόψη μας. Η ενεργειακή απόδοση είναι καθοριστική ζωτική σημασία για τα κτίρια, τι υποδομέ, τι μεταφορέ, την τεχνολογία, τι επικοινωνίε. Όλοι αυτοί οι τομεί και πολλοί άλλοι κλάδοι εξαρτώνται από την ενεργειακή απόδοση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συντονισμένε και διαρθρωμένε πολιτικέ, γιατί αλλιώ θα πετύχουμε του στόχου μα. Η ενεργειακή απόδοση είναι θεμελιώδης επίσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όπως αναφέρθηκε, λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα μείωση των εκπομπών. Δεν μπορούμε να κάνουμε παράλληλες συζητήσεις, άλλα να λέμε για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλα για την ενεργειακή απόδοση. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε κάποια σημεία που θεωρώ καθοριστικά. Πρώτον, είναι σημαντικό να υπάρξουν δεσμευτικοί στόχοι. Το να μιλούμε για εθελοντικά, για θελούσια κριτήρια, Μάλλον τα εθελούσια κριτήρια είναι αυτά που μας έφεραν στην κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεσμευτικούς στόχους γιατί δεν θα έχουμε το 20%. Τι μήνυμα όμως περνάμε με τον τρόπο αυτό στους πολίτες. Ότι στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Διότι έχουμε έναν στόχο που το πολύ πολύ να φτάσει το 9%. Και δεν θα πετύχουμε το 20% μείωσης γιατί δεν υπήρχαν δεσμευτικοί στόχοι. Οι δεσμευτικοί στόχοι είναι αυτοί που επιτρέπουν και παροτρύνουν υλοποίηση των πολιτικών. Δυστυχώς ε, χρειάζεται να προσφύγουμε μόνο σε πολιτική βούληση, σε καμία άλλη κατηγορία βουλήσεων, βουλήσεως. Η τύχη του στόχου αυτού θα μας επέτρεπε να δημιουργήσουμε ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Κάτι που δεν είναι αμεληταίο αυτή την εποχή. Αυτό που βλέπουμε εδώ, το βλέπουμε και στην οικονομική πολιτική της Ένωσης. Δεν είναι σε θέση η Ένωση να δημιουργήσει μια κοινή πολιτική για τη δημιουργία θέσεων νέων θέσεων εργασίας. Δεν είναι ικανή επίσης να προχωρήσει στην ενεργειακή απόδοση. Ελπίζω στον τομέα των κτηρίων τουλάχιστον να μπορέσουμε να δώσουμε μια συντονισμένη απάντηση αύριο που θα είναι και απάντηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Τελευταίος αγωγητής εξ ονόματος των ομάδων, ο κύριος Πάσκα. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η επεξεργασία του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση περιγράφει πολλές δυνατότητες για το πόσο μπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου το 2020. Η βασική σκέψη αυτού του εγγράφου βασίζεται στην ε, εξής λογική. Θα πρέπει να έχουμε μια ορθολογική διαχείριση της ε, ενέργειας σε διάφορους τομείς όπου θα πρέπει να ληφθούν αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια εξοικονόμηση ενέργειας και να μειώσουμε και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Τα πρωταθέντα μέτρα στο τομέα των ενεργειακών υποδομών της παραγωγής ενέργειας και της μεταφοράς της κλπ. Και όλα αυτά τα μέτρα όμως περιγράφονται γενικά, χωρίς να περιγράφεται ακριβώ η χρησιμότητα αυτών των μέτρων. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έναν κατάλογο των αναγκαίων μέτρων, ούτως ώστε να μπορεί να αυξηθεί η βαθμία ενεργειακή αποδοτικότητα. Εν ώψη του στόχου του 2020 της ε, μείωσης ε, κατά 20% θεωρώ ότι θα είχε νόημα να δούμε ποια μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ποιο βαθμό, με ποιο κόστος και με ποια χρησιμότητα. Και μάλιστα τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν ε, ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το στόχο της ενεργειακής αποδοτικότητας όσον αφορά την παραγωγή και μεταφορά της ενέργειας. Αλλά όσον αφορά το, αλλά σε σχέση με το υψηλό κόστος έχω δυστυχώς την άποψη ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα μέχρι το 2020. Γι' αυτό έχω την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί επιλεκτικά όσον αφορά την οργάνωση, τον χρόνο και τα, την οικονομική ε, ε, και τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων ούτω ώστε να δοθεί μια όφηση καταρχήν στους επιρρογνώμονες και στη συνέχεια στο ε, επίπεδο της ε, κοινή ε, γνώμης. Στον τομέα της μόνωσης, στον τομέα των οχημάτων και των ηλεκτρικών συσκευών μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα ώστε οι καταναλωτές να αγοράζουν συσκευές για παράδειγμα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος για να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρινς. Δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μία ερώτηση. Ποιος γνωρίζει πόσο πετρέλαιο και αέριο εισάγουμε στην Ευρώπη. Ποιος γνωρίζει πόσες ποσότητες αυτών των πόρων υπάρχουν στην Ευρώπη. Η απάντηση είναι δεν έχουμε πολλούς τέτοιους ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη και χρειάζεται να εισάγουμε τεράστιες ποσότητες αερίου και πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και την Ρωσία. Αυτή η εξάρτηση από τις εισαγωγές αυξάνεται και είναι, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δημιουργήσουμε σχέσεις, να αναπτύξουμε σχέσεις με τρίτες χώρες. Ας σκεφτούμε για λίγο αγαπητοί συνάδελφοι. Τι σημαίνει εισαγωγή αερίου πετρελαίου για τους πολίτες μας. Σημαίνει ότι εξάγουμε <clears throat> χρήμα ευρωπαϊκό σε αυτές τις τρίτες χώρες. Εξάγουμε το χρήμα μας για να εισάγουμε πετρέλαιο και αέριο. Τι ξέρουμε για το μέλλον. Ξέρουμε ότι στο μέλλον το πετρέλαιο και το αέριο, η τιμή του πετρελαίου και του αερίου θα αυξηθεί διότι αυτοί οι πόροι θα γίνονται όλο και πιο σπάνιοι. Με αποτέλεσμα στο μέλλον, αν δεν αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο κατανάλωσής μας, θα, εξακολουθούμε, θα εξακολουθήσουμε να εξάγουμε το χρήμα εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει ένας απλός τρόπος όμως πώς να σταματήσουμε αυτή τη μαζική εξαγωγή χρήματος. Ένας πολύ απλός τρόπος. Πρέπει να εξοικονομούμε ενέργεια, πρέπει να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση. Εξοικονομώντας ενέργεια θα εξοικονομήσουμε και χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να επενδύσουμε όχι στις τρίτες χώρες αλλά στις δικές μας οικονομίες. Καλό λοιπόν όλους μας να υποστηρίξουμε την έκθεση του κυρίου Μπένσεν για την ενεργειακή απόδοση διότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις εθνικές μας οικονομίες. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η κυρία Ούλσκοφ έχει το λόγο. Πρόεδρε, και εγώ ξεκινώ ευχαριστώντας ε, τον εισηγητή για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε στην σαφέστατη έκθεσή του. Πρέπει να έχουμε το συντομότερο δυνατό δεσμευτικού στόχου ενεργειακή απόδοση για πολλούς λόγους. Οικονομικούς, ανταγωνιστικότητας, θέσεων εργασία, προστασία του κλίματο. Ο κύριο Έτιγκερ μίλησε για την ενεργειακή εξοικονόμηση και τη διαφορά της από την ενεργειακή απόδοση. Αλλά περί πρόκειται. Στη χώρα μου λέμε ότι ότι είναι, περιττό ανά, ότι είναι κακό να ανάβεις περιτά μια φωτιά, ότι δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιείς ε, χωρίς λόγο τους πόρους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ε, εξισορρόπηση μεταξύ της παραγωγής ενέργειας και της κατανάλωσής της. Οπότε για να υπάρχει μια καλύτερη, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρέπει να έχουμε έξυπνο τρόπο χρησιμοποίησης της ενέργειας. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους ε, έχουμε κοινούς στόχους, αλλά πρώτα πρέπει να βρούμε μια συμφωνία για κοινέ μετρήσει και κατόπιν να αποφασίσουμε επί δεσμευτικών στόχων. Εμείς αυτή τη στιγμή αξιολογούμε την ε, τις συνέπειες της μη ύπαρξης δεσμευτικών στόχων. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει μια αλλαγή στο μέλλον και υποστηρίζουμε λοιπόν την έκθεση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ζητούσα από τους συναδέλφους να τηρούν το χρόνο που τους έχει δοθεί. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή απόδοση ήταν πάντα ο σημαντικότερος πόρος ο γίγαντας που κοιμάται και εδώ κρύβεται ένα τεράστιο δυναμικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ωραίο εδώ είναι ότι αυτό είναι απογυμνωμένο από ιδεολογίες. Μπορεί κανείς να προσεγγίσει το θέμα από μια ουδέτερη άποψη. Το μόνο το οποίο μα διχάζει είναι το ζήτημα τη δεσμευτικότητα των στόχων. Κύριε Πίτρο, θα πρέπει να πάω, μου αρέσει η προσέγγιση σα για τι δύο βαθμίδε, τα δύο στάδια. Ότι καταρχήν να δείξουμε εμπιστοσύνη προ τι χώρε μέλη και καταρχήν να θέσουμε το ζήτημα σε θελούσιες συμφωνίες. Και αν διαπιστώσουμε ότι οι στόχοι μέχρι το 2020 δεν έχουν τηρηθεί, τότε ίσω να προχωρήσουμε σε δεσμευτικού στόχου. Νομίζω ότι η έκθεση πηγαίνει προ την ορθή κατεύθυνση δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική. Θα ήθελα να τονίσω μόνο ένα θέμα, το θέμα των περιφερειακών ταμείων. Αναφέρθηκα σε αυτό κύριε Επίτροπε. Με τα περιφερειακά ταμεία και τα ταμεία συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο δεν αξιοποιούμε παρκώ. Και εδώ στο τομέα τη ενεργειακή απόδοση θα μπορούσαμε επιτέλου να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή υπεραξία την οποία εφαρμόζουμε αποτελεσματικά με καινοτόμο τρόπο. Κάτι το οποίο δεν πράξαμε στο παρελθόν και εγώ ω εισηγητή για την απαλλαγή του προπολογισμού τη Επιτροπή, βλέπουμε πόσα χρήματα σπαταλήθηκαν στο μέτρο της συνοχής. Ας πάψει αυτή η κατάσταση. Θεωρώ πολύ καλό κύριε Επίτροπε ότι εδώ βάζετε μια προτεραιότητα λέγοντα ότι τα ταμεία αυτά θα πρέπει να εξοπλιστούν καλύτερα για το θέμα τη ενεργικής απόδοση γιατί μόνο έτσι θα κατορθώσουμε πράγματι να επιτευχθεί μια συνοχή τουλάχιστον στον ενεργειακό τομέα. Αλλά θα ήθελα να σα προειδοποιήσω για το εξή. Για, φανατισ... Ε, για ε, προπαγάνδες όπως αυτές που είδαμε με το τηλέφωνο του ντους ε, πράγματα που φοβίζουν ε, τους πολίτες θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση στον αφορά την ενεργειακή απόδοση θα έχουμε αυτό το στόχο κατά νου χωρίς όμως τέτοιου είδους φανατικές εκστρατείες που τελικά έχουν σαν αποτέλεσμα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποθαρρύνονται Ευχαριστώ πολύ Και εγώ ευχαριστώ Κύριε Σέικχαουτ, δύο λεπτά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βέντσον για την εισήγησή του, για την έκθεσή του, διότι νομίζω ότι μας άνοιξε το δρόμο για τα επόμενα χρόνια. Βεβαίω θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στην κατάλληλη προοπτική. Το 2050, 15 συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει περιορίσει τις κατα... 90-95% της ε, εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, οπότε θα χρειάζεται και να εισάγουμε λιγότερες ποσότητες. Και δεν θα χρειάζεται να αναπτύξουμε και να αξιοποιήσουμε άλλες ε, μορφές και πηγές ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, λένε, δεν επαρκούν για να πετύχουμε το στόχο μας. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε ορισμένους συγκεκριμένους τομείς. Καλύτερη μόνωση των κτηρίων, παραδείγματος χάρη. Αν ρίξουμε μια ματιά στο περιβάλλον, αντιλαμβανόμαστε ότι 5% της ενέργειας που καταναλώνεται από το περιβάλλον για διάφορους σκοπούς και το 40% της κατανάλωσης προέρχεται από τα κτίρια. Θα χρειαστούμε λοιπόν πάνω από 60 χρόνια για να ανανεώσουμε και να ε, ε, βελτιώσουμε τη μόνωση όλων των κτιρίων που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα, τη καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Αυτή θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα, αν εφαρμοστεί, αν γίνει σωστά, αν γίνει σωστά θα φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα και δεν θα χρειάζεται να εισάγουμε ενέργεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζιόμπρο, δύο λεπτά. Πρόεδρε. Το Σεπτέμβριο του 2009 στην Ευρώπη αρχίσαμε να αντικαθιστούμε παραδοσιακούς λαμπτήρες με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Και αυτό έγινε για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Ε, και παρόλο που ήταν πολύ ψηλό το κόστος αυτής της αντικατάστασης για τον πολίτη σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα ε, και είναι ένα, δεν ξέρω αν είναι μυστικό ότι τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχθησαν από διαφημιστικό υλικό των κατασκευαστών αυτών των ηλεκτρικών ε, λαμπτήρων οικονομίας. Ε, νομίζω ότι δεν λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη τις ε, διαφορές μεταξύ των χωρών καθώς και το κόστος το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί αν εφαρμοστούν αυτές οι οδηγίες. Ε, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου θα είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Ο κύριος η αναζήτηση της οικονομίας είναι μία πρόκληση για να μειώσουμε την εξάρτηση από άλλες πηγές, για να έχουμε πιο χρήματα στα διάθεσή μας, για να αξιοποιήσουμε άλλες πηγές ενέργειας και να αναζωογονήσουμε τις ε, διάφορες περιοχές, τις και τις περιφέρειές μας. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στις ε, εργατικές και κοινωνικές κατοικίες. Πρέπει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτό το σκάνδαλο που επιβάλλει στους φτωχότερους την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ οι πλουσιότεροι έχουν τη δυνατότητα με διάφορους τρόπους να μειώνουν, να ε, χρησιμοποιούν όλη την ενέργεια που χρειάζονται χωρίς να πληρώνουν το πλήρες κόστος. Πρέπει να γίνονται οικονομίες παντού, όπως γινόταν στη Γαλλία, προτού να επέμβουν οι γαλλικές οδηγίες για την ενιαία αγορά ενέργειας. Ένα από τα πρώτα μέτρα θα ήταν να διασπάσουμε την ενιαία αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα προϊόν όπως η ηλεκτρική ενέργεια που δεν αποθηκεύεται και μεταφέρεται δύσκολα είναι κάτι το παντελώ τρελό. Η ενεργειακή απόδοση θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ποιότητα αν στηριχθεί σε μια στρατηγική ενεργειακή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση που θα ξεφύγει από του περιορισμού τη ελεύθερη αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτσιν Δύο λεπτά. Πρόεδρε, πιστεύω ότι όντως πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων έξυπνων συστημάτων μέτρησης που θα επιτρέπουν να μετρούμε την εξοικονόμηση γενέργειας. Τούτο πρέπει να γίνει και από πλευράς διανομέων και από πλευράς κατασκευαστών. Όλοι οι κλάδοι πρέπει να εμπλακούν και γιατί θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης κάτι τέτοιο. Αν δίνουμε άδειε για νέες υποδομές θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την ενεργειακή απόδοση αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας που προσφέρουν οι υποδομές αυτές. Πιστεύω ότι τούτο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και για την Ουγγρική και για την Πολωνική Προεδρίας. διότι θεωρώ ότι το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας θα επιτρέψει την υιοθέτηση μιας σειράς πρωτοβουλειών νομοθετικών ή όχι για να έχουμε έναν πιο ε, αποτελεσματικό ευρωπαϊ... μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική ενεργειακής απόδοσης. Μετά το Κανκούν αναρωτιέμαι μπορούμε να κάνει κανεί... μπορεί να κάνει κανείς ρεαλιστικές προβλέψεις για την αλλαγή του κλίματος. Πιστεύω πάντως ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση και να αναθεωρήσουμε την προσέγγιση μας στην, στην κατανάλωση ενέργειας ε, στην Ένωση. Ένα δε θέμα κλειδί είναι οι μεταφορές για να έχουμε πιο αποτελεσματική ενεργειακή απόδοση. Στοχεύοντας ε, με έμφαση στη μείωση της ζήτησης και εδώ πρέπει να αναλάβουμε δράση έναντι των πολιτών. Προφανώς όλα αυτά θα είναι θετικά και για τον πολίτη και για τον καταναλωτή και για τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεάντζελης έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του συναδέλφου Μπένσεν είναι θετική για τέσσερις τουλάχιστον λόγους. Ένα, επαναλαμβάνει ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος μείωση των εκπομπών που αλλάζουν το κλίμα και ότι μια επένδυση ε, στον τομέα αυτό θα οδηγήσει και οικονομική αύξηση και θέσεις εργασίας διότι παρέχει σωστές προτάσεις για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και διότι καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει με αποφασιστικότητα στην επαγγελματική κατάρτιση, την πρόσβαση στην ενημέρωση της μικρομεσαίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αναδιάρθρωση και την αναμόρφωση των υφισταμένων κτηρίων. Διότι προτείνει συγκεκριμένους στόχους, διότι επιβεβαιώνει το εργαλείο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, βάσει της οποίας ε, αγοράζονται εγγυημένες ε, εξοικονομήσεις με ε, δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση των, του κόστους του ηλεκτρισμού για τον πολίτη. Η έκθεση θα είναι ακόμα πιο χρήσιμη αν κατορθώσει να καθορίσει ξεκάθαρα δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές. Θα πρέπει το στόχο του 20% να τον υλοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε τις ευκαιρίες αυτής. Θα ήταν ένα, κάτι θα ήταν ένα θαρρυντικό μήνυμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτοφ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι Η υψηλή ενεργειακή απόδοση είναι σημαντικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον απαραίτητο στοιχείο της ε, ε, στρατηγικής για μια ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη απασχόληση και σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα. Η ψηφοφορία για το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση θα μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη για ε, ταχεία, ταχεία, ταχείες επεμβάσεις. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια εκτεταμένη ανάλυση της νομοθεσίας που υπάρχει για αυτό τον τομέα η ανακαίνιση των νέων κτηρίων και υψηλότερα κατασκευαστικά πρότυπα, πιο αποτελεσματικές υποδομές, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και των οχημάτων είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που θα για την ενεργειακή απόδοση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 η ενεργειακή απόδοση πρέπει να φέρει οικονομικά ωφέλη και πρέπει να συμβάλλει στο δημόσιο καλό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιγκερέντο. Η κυρία Φιγκερέντο, συγγνώμη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι απαραίτητο να προβούμε σε μία αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για το 2017. Να διαφοροποιήσουμε τα μέσα για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης. Το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης δεν μπορούμε να το επικαλούμαστε για να μην πετύχουμε το στόχο της μείωσης του κατά 20% μέχρι το 2020 είναι απαραίτητο να βρεθεί μια λύση για το πρόβλημα της ενεργειακής ένδυας ή παινίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κίνα και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και πρέπει να προβλέψουμε τη χρηματοδότηση μέτρων που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, των μεταφορών, των ε, ε, κοινωνικών κατοικιών κλπ πρέπει να εξασφαλίσουμε τις αναγκαίες πιστώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τις οικογένειες και τις χώρες που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα. Η ενεργειακή, απόδοση δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα κύριος κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάσετε ένα πολύ καλό σχέδιο και νομίζω ότι ο συνάδελφος κύριος Μπέντσεν ε, το βελτίωσε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να πετύχουμε ε, την, την ε, περισσότερη μεγέθυνση με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε πιο, ενεργ προϊόντα τα οποία να είναι σχεδιασμένα βάσει τη ενεργειακή απόδοση. Αλλά θα πρέπει επίση να μειώσουμε και του λογαριασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο. και θα πρέπει να βρούμε καινοτόμε λύσει και τα σωστά πολιτικά κίνητρα. Πάντοτε αποδεικνύεται στην ιστορία τη οικονομία, ότι εκείνε οι οικονομίε ήταν πιο αποτελεσματικέ που πέτυχαν την ε, απόδοση είτε στον τομέα πρώτων υλών είτε στον τομέα της ενέργειας. Και εμείς οι Ευρωπαίοι με το υψηλό επίπεδο ζωής ε, εδώ καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Θα πρέπει να πετύχουμε επίσης τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους και να μειώσουμε την εξάρτηση από τις ορυκτές πηγές ενέργειας. Βεβαίως, ε, ε, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό ενέργειας. Ε, θεωρώ ότι αυτό που είπατε ότι δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτική στόχη, είναι σωστό. Δεν θα πρέπει νομίζω να χανόμαστε μέσα σε, σε συζητήσεις σχετικά με τους ορισμούς της ενέργειας. Θεωρώ ότι η Κομισιόν και ο Συγητής υπέδειξαν τον ορθό δρόμο το ότι οι στόχοι δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι. Οι στόχοι θα πρέπει να παραμείνουν φιλόδοξοι και αυτό για εύλογους ε, λόγους. Γι' αυτό η πολιτική μας ε, ομάδα θα το καταψηφίσει. Ο κύριος Βόμποντα έχει το λόγο. Ε, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Μπέντσεν για την πολύ καλή του έκθεση. Μόνο που θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, κύριε Επίτροπε. Προέρχεστε από το χώρο τη περιφερειακή πολιτική και από ένα σημαντικό ομόσπονδο κρατήδιο τη Γερμανία. Εγώ προέρχομαι από την περιφερειακή πολιτική δεν θα πετύχουμε μη δεσμευτικού στόχου εάν δεν ε, κερδίσουμε τους Δήμους και τις ε, περιφέρειες και δεν τοποθετούμε σε αυτό το περιφερειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, η πολιτική μεταφορών, τα μεταραξυγένσεις, η καταπολέμηση ενεργικής πενίας. Όλα αυτά δεν ρυθμίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο των πόλεων. Γι' αυτό θα πρέπει εδώ να επικεντρώσουμε την προσοχή μα. Θα πρέπει να κερδίσουμε του Δήμου και τι κοινότητε για ένα μείζον ευρωπαϊκό εγχείρημα τη ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργεια. Ε, θα ήθελα να σας καλέσω εδώ να ε, κάνετε κάποιους προβληματισμούς σχέση με το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε περισσότερο τον πολίτη ακριβώς μέσω των δήμων, των περιφερειών και των κοινοτήτων. Γιατί αυτή τη σύνδεση είναι σημαντική, ούτω ώστε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους της αύξησης ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καρβά... Η κυρία Καρβάλιο, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Κύριε Επίτροπε, η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτική σημασία αν θέλουμε να αυξήσουμε τον ενεργειακό εφοδιασμό μας, να περιορίσουμε τι εκπομπέ αερίου θερμοκηπίου και να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ενταγωστικότητα των κοινωνιών μα. Η ενεργειακή απόδοση σημαίνει να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα μέσα, με λιγότερου πόρους. Η έκθεση μα παρουσιάζει μια φιλόδοξη προοπτική για την επίτευξη αυτού του στόχου χάρη στην εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων και θετικών κινήτρων. προβλέπονται σημαντικά μέτρα για τον εξυγχρονισμό της τεχνολογίας, τα έξυπνα, τα εφή δίκτυα δηλαδή. Μέτρα επίσης σε ό,τι αφορά το τομέα των κατασκευών, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των μεταφορών. Σκοπός είναι να διπλασιαστούν οι πόροι για την τεχνολογική ανάπτυξη και την τεχνολογική έρευνα και για τα σχέδια επίδειξης στον ενεργειακό τομέα η έκθεση επιμένει στην ανάγκη των διαφορετικών ταμείων για να, φτάσουμε σε μια καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τον προϋπολογισμό της, κοινο... της Ένωσης μετά το 2013. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Μπέντσεν για τη θαυμάσια δουλειά που έκανε για την ισορροπία που κατάφερε να βρει και καλό όλους τους βουλευτές να υποστηρίξουν και να υπερψηφίσουν αυτή τη σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Καρβάλιο. Ο κύριος Μπαρτσίδης έρχεται. Θα λάβει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, επίτροπε, παρότι η ενεργειακή απόδοση έχει εμφανιστεί σε πολλά νομοθετικά κείμενα, τα αποτελέσματα είναι, είναι ξεκάθαρα. Ούτε το μισό του στόχου των 20% δεν θα πετύχουμε. Το ενδεύτερο δηλαδή. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα. Η Επιτροπή καλά κάνει και αναθεωρεί το πρόγραμμα δράση έπρεπε να λάβει υπόψη ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν επαρκώς τα μέτρα εξοικονόμησης για να αυξήσουν και την ενεργειακή ασφάλειά τους. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν δεσμευτικοί στόχοι στα κρατημέλη για την ενεργειακή απόδοση, στόχοι που θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται. Είδε μη, δεν θα υλοποιήσουμε τους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι έχει το λόγο δύο λεπτά. Πρόεδρε, Είμαι πολύ ευτυχής που παίρνω το λόγο για αυτή την έκθεση, η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική, διότι μιλάμε για τους στόχους της μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά παράλληλα νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ως οικονομίες, προστατεύοντας, ενώ θα προστατεύουμε το περιβάλλον και το πορτοφόλι των πολιτών σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια δράσης, υπάρχει περιθώριο ελιγμού για τη βελτίωσή τους. Πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε σε δύο φάσεις. Πρώτα σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη και αν δεν καταφέρουμε τίποτε τότε θα πρέπει να παρεμβούμε πιο δυναμικά. Έχω συζητήσει το θέμα με συναδέλφους και πολλοί συμφωνούν μαζί μου και απευθύνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε τα αναγκαία μέσα για να εξασφαλίσετε την τήρηση, το σεβασμό της νομοθεσίας. Εάν χρειαστεί να είσαστε πιο αυστηροί θα μπορέσετε να προβείτε σε αναλύσεις και να μας δώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Τα διορθωτικά ταμεία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν. Τα κονδύλια που είναι διαθέσιμα ποτέ, ποτέ, ποτέ, σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούνται για έργα ενεργειακής απόδοσης. Γι' αυτό κατέθεσα για το άρθρο 81 μια τροπολογία. Μια τροπολογία που έχει σκοπό να διευκρινίσει περισσότερο το κείμενο. Δεν χρειά... Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και όπως είπε και ο κύριος Βόμποντα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η τοπική και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να εμπλακούν περισσότερο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μπορούμε να, ε, ακόμα, επίσης και οι πολίτες πρέπει και αυτοί να συμμετάσχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Στην Ολλανδία υπογράψαμε μια σύμβαση με τη βιομηχανία με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστική μείωση κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Τικάου. Πρόεδρε, Επίτροπη. Πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες έχουν υφίστανται την ενεργειακή παινία. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι πολιτικές προστασία της ενεργειακής απόδοσης. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι τα οι εργατικέ κατοικίε. Μόνο το 1% των κτηρίων του 2020 θα είναι καινούργια. Άρα, ε, εφόσον μιλούμε για δεσμευτικούς στόχους ε, στα υφιστάμενα κτίρια, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε και για χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν λοιπόν μια σειρά φορολογικών κινήτρων που θα προωθούν την ενεργειακή απόδοση. Πρόσφατα στο Κοινοβούλιο είχαμε μια ε, συνάντηση ε, για την, ε, μια εκδήλωση για, την, για τα πέντε χρόνια της ύπαρξης αυτής της πρωτοβουλίας. Ωστόσο, πολλοί από τους παρόντες εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης δεν ήξεραν καν την πρωτοβουλία για την ενεργειακή απόδοση. Το ποσό θα έπρεπε πολύ μικρό ποσό από το τα περιφερειακά ταμεία πηγαίνουν στην ενεργειακή αποδοχή των κτηρίων. Ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε να χρησιμοποιήσετε την ενδιάμεση αξιολόγηση για να δώσετε μεγαλύτερα, περισσότερα κονδύλια σε προγράμματα ενεργειακής απόδοση και για να αυξήσετε τι δυνατότητε χρήση έως και 15% του Περιφερειακού Ταμείου στα, ε, σε τέτοια έργα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος Καντσιάν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κύριο Μπένσεν, που ήταν πολύ σωστό στην έκθεσή του. Ο Επίτροπος ξεκίνησε τη συνεδρίαση λέγοντας ότι και συμφωνώ μαζί του ότι το να μιλάμε σήμερα για απόδοση ε, το κάνει είναι μια πολύ θεωρητική ε, συζήτηση. Ήδη μιλάμε για το ενδεύτερο του 20%, όχι για το 20%. Προσθέτει ότι πρέπει να ενισχυθεί η κουλτούρα της εξοικονόμησης. Μιλούμε για ένα κλίμα, για μια χρονική στιγμή που πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Πώς? Πιστεύω ότι πρέπει καταρχάς να προχωρήσουμε προς την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Και για τα κτίρια άρα την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και ιδίως την ενεργειακή απόδοση των μεταφορών. Θα ήθελα να σταθώ για λίγο στο πολύ σημαντικό γεγονός των κατάλληλων πόρων για την επίτευξη των στόχων που, έθεσα, που θέτουμε πιστεύω ότι πρέπει να δαπανίσουμε για να εξοικονομήσουμε. Έλεγε σήμερα ο κ. Μπαρόζο στη, στην Ολομελία ότι δεν θα περάσουν τα ευρωομόλογα και έλεγε ότι έχει τη δυνα... υπάρχει δυνατότητα νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Κύριε Επίτροπε, εμείς πριν από λίγο καιρό ξεκινήσαμε πρόσφατα εγκρίναμε μία έκθεση για τη θέση της ενός ταμείου που λαμβάνει υπόψη τα παλιά προγράμματα αποκατα... Ε, ε, ανάκαμψης για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων εξοικονόμησης. Αυτό θα ήταν καθοριστικό και συμβολικό ακόμα για να θεσπιστεί μια αρχή, να προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο σε μια λογική ΣΔΙΤ, εξορθολογικοποιώντας τα, τα κονδύλια που έχουμε και από το Ταμείο Συνοχής και από αλλού, ε, με τρόπο που θα προσελκύει η Ευρώπη και δεν θα δίνει μόνο ε, κονδύλια δωρεάν, χρησιμοποιώντας καλύτερα τους υφιστάμενους πόρους και δίνοντας πραγματική σημασία στα αποτελέσματα. Αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό σύστημα για να προχωρήσουμε στην αναζήτηση πόρων και να επιτρέψουμε να μην είναι πλέον ταμπού η εξοικονόμηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίλο έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε επίτροπε, συνάδελφοι. Η αναθεώρηση του προγράμματος δράσης για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση που επιτρέπει να ε, συμπεριλάβουμε τις διάφορες στρατηγικές της Ευρώπης. Αν ε, επενδύουμε στην ενεργειακή απόδοση από τη μια μεριά και αυτό είναι θεμελιώδες γιατί συμβάλλει στην επίτευξη το 2020 των στόχων μείωσης των εκπομπών από την άλλη ωστόσο είναι σκόπιμο να μείνουμε στις πρωτοβουλίες εκείνες που επιτρέπουν καλύτερη εκμετάλλευση της εξοικονόμησης ενέργειας στην Ένωση που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται. Είμαι ικανοποιημένος διότι μεγάλο τμήμα αφιερώνεται στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Προς την κατεύθυνση εκείνη πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιχειρήσεις μας θα πρέπει να επανεξετάσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο το κατά πόσον τόσο τις παραγωγικές διεργασίες όσο και τα προϊόντα τους είναι σημαντικό να υπάρξουν στόχοι απο... ε, ε, ε, δεσμευτικοί στόχοι απόδοση χωρίς τους οποίους δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο μας στην Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτά. Τελευταίος η κυρία Ποδηματά. Κύριε Πίτροπε, θέλω να επιμείνω σε ένα σημείο στη σημασία που έχει η θέσπιση ενός δεσμευτικού στόχου ενεργειακής αποδοτικότητας για την ευρωπαϊκή οικονομία σε συνθήκες δύσκολες οικονομικές για μια σειρά κράτη μέλη που χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη για την προστασία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ένας δεσμευτικός στόχος θα δημιουργήσει το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού δυναμικού ευρωπαϊκών εταιριών κυρίως μικρομεσαίων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες και στις υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας. τα κράτη μέλη θα αποκτήσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να ενισχύσουν εκείνες τις αγορές που σε κάθε οικονομία μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσει εργασία. και επιπλέον θα υπάρχουν σημαντικά συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη για τα νοικοκυριά για τι επιχειρήσει, για το δημόσιο καθώ θα απολαμβάνουν χαμηλότερου λογαριασμού ενέργεια. θέλω λοιπόν να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του και να καλέσω την ευρωπαϊκή επιτροπή να υλοποιήσει τι προτάσει τη έκθεση μπεντσεν διευκολύνοντα παράλληλα την έξοδο τη οικονομία μα από την κρίση. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω παρακαλώ να τηρείτε τον χρόνο που σας έχει δοθεί. Προχωρούμε τώρα στη ε, διαδικασία Catch the Eye. Δυστυχώς δεν θα δώσω το λόγο σε όλους όσοι το ζήτησαν. Θα χρησιμοποιήσουμε στόσο τα πέντε λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτος, ο κύριος Πέτερ Ιάρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, φυσικά η ενεργειακή απόδοση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολύ οικονόμοι όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή τις ορυκτές πρώτες αλλά θα πρέπει, όμως, να είμαστε ρεαλιστές ε, και θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και για την ε, κοινωνία και για τον πολίτη όταν ορίζουμε κάποια ποσοστά. Και θα πρέπει όλα αυτά να μπορεί να τα πληρώσει και ο πολίτης. Επίσης ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να τα κατανοεί όλα αυτά. Γιατί αν δεν υπάρχει αποδοχή στο πληθυσμό δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Και ακριβώς αυτή είναι η πτυχή που θεωρώ ότι παραμελείται στην λόγω έκθεση. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε τον χρόνο μιλίας και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αρσένη. Οι διαπραγματεύσει στο Κακούν ε, σημείωσαν σχετική επιτυχία. Οι διαπραγματεύσει για την κλιματική αλλαγή προχωράνε. Ε, χώρες όπως η Κίνα δεν περίμεναν ε, το αποτέλεσμα στο Κακούν. Παίρνουν μέτρα ε, ακόμα και ε, το διάστημα μετά την αποτυχία της Κοπεχάγης. Αν δεν επενδύσουμε και εμείς σε θέματα όπως είναι η ενεργειακή απόδοση και η ενεργειακή εξοικονόμηση, τότε θα χάσουμε διπλά. Από τη μία, τα νοικοκυριά μας, οι επιχειρήσεις μας, οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να πληρώνουν παράλογα κόστη. Από την άλλη, θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε την πράσινη πρωτοπορία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι άμα σήμερα δυσκολευόμαστε να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η κίνα πώς θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε στο μέλλον μια πράσινη κίνα. γι' αυτό είναι πραγματικά σημαντικό να υποστηρίξουμε και να λάβει η ευρωπαϊκή ένωση ένα δεσμευτικό στόχο για τη μείωση της ε, ενεργειακής για ενεργειακή εξοικονόμηση στο. 20%. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ. Με την πολιτική ενεργειακής απόδοσης ε, όπως ξεκινούνται τώρα από τα κράτη-μέλη, θα πετύχουμε τον στόχο του 20% το 2020 για μείωση της ενεργειακής ε, απόδοσης, ένα, ούτε καν 10% από το κοντευτικό αποτέλεσμα. Αν αυξηθεί η ενεργειακή κατανάλωση θα τεχθεί σε κίνδυνο και η επίτευξη του στόχου του 20% για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, γιατί ο στόχος αυτός βασίζεται στο, στην τελική κατανάλωση της Ένωση, με υπέρ δεσμευτικών στόχων και στην ενεργειακή απόδοση για να εξασφαλίσουμε ότι οι ενεργειακέ πολιτικέ πιο αργά παρακαλώ, λέει ο ενισχύονται. Δυστυχώς, το να στηριζόμαστε στην καλή προαίρεση των κρατών μελών δεν αποτελεί θετική στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να χαράξει το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθηθεί με στόχου ε, πολιτική σαφού και αποτελεσματικού. Να σταματήσουμε να επενδύουμε. Θα πρέπει να επενδύουμε σε νέε δομέ παραγωγή ενέργεια ε, που, να που μπορούμε εκτός ε, από την ε, καθαρή ενέργεια να μειώσουμε την ενέργεια. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία το 2011 για την ενεργειακή απόδοση των υφισταμένων κτίριων. Αυτό είναι καθοριστικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ενεργειακή απόδοση είναι λέξη κλειδί για την οικονομία του μέλλοντος δεν πρέπει να, επιβάλλεται ωστόσο, αλλά να ενθαρρύνεται. Χρειάζεται να παρέμβουμε έναν των κρατών μελών, ούτω ώστε όποιο επιλέγει τη βελτίωση τη της απόδοση επιχείρηση ή τη κατοικία του να λάβει κίνητρα. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ε, ιδιώτε να επενδύσουν χωρί να του πείσουμε ή να του ενθαρρύνουμε. Η βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση σημαίνει να βοηθούμε το περιβάλλον, να εξοικονομούμε ενέργειε. Είναι ωστόσο θεμελιώδο να συνδέσουμε τι επιλογέ αυτέ σε ένα τόσο λεπτό ε, πεδίο με ευρωπαϊκές πολιτικές που στοχεύουν στην δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Οι δεσμευτικοί στόχοι ε, περιλαμβάνουν περιτές και συχνά ε, αλυσιτελείς δαπάνες, ενώ δεν πείθουν τους πολίτες ότι η εξοικονόμηση στον τομέα αυτό σημαίνει ότι εξοικονομούμε και στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγκεντη έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κατά την άποψή μας, οι, οι, τη της, οι αιτίε της κλιματικής αλλαγής ε, δεν ε, συνδέονται με το, δεν άγονται μόνο στον άνθρωπο. Βεβαίω είναι δική μας ευθύνη να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε τις ε, κλιματικές ε, μεταβολές και να αποκαταστήσουμε την πρωταρχική κατάσταση της ε, φύσης. 4% της ενεργειακής κατανάλωσης στον κόσμο 40% μάλλον καταναλώνονται για την κατασκευή κτηρίων. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν ε, την κατασκευή νέων ε, κτηρίων και θα πρέπει να ανακαινήσουμε τα παλαιά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειώσουμε την ε, κατανάλωση ενέργειας από τα αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας νέες υβριδικές τεχνολογίες και νομίζω ότι θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες να στραφούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπατσέσκου, ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, θα ήθελα να τονίσω ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι φέρνει ουσιαστικά οικονομικά ωφέλη αλλά και κοινωνικά ωφέλη όπως δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέχρι το 2020 η ανάπτυξη και εμπορία νέας προηγμένης τεχνολογίας είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό οι ενεργειοβόρες ε, επιχειρήσεις πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικές στα πλαίσια της, του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να προωθούμε την επίτευξη των ε, ενεργειακών στόχων Θέλω να συγχαρώ τις προσπάθειες Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ενιαίου ενεργειακού δικτύου. Περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης για τα έργα υποδομής. Ευχαριστώ. Ωραία. Η κυρία Στάιλ τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μπένσεν που αναφέρθηκε στην κατασκευαστική βιομηχανία. Η έκθεσή μου για την κατασκευαστική βιομηχανία, στα πλαίσια αυτής της έκθεσης συζητήσαμε το θέμα της ενέργειας. Ο κύριος Βόμποντα αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλω να ε, πω πόσο ότι ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, είχαμε περικοπές των κονδυλίων που πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μιλάμε για έξυπνους, αναφέρονται οι έξυπνοι μετρητές στην έκθεση και θα μπορέσουμε να πετύχουμε το, το στόχο, ε, κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει κανείς πάνω από την Προεδρία, το στόχο της ε, ε, ευρείας χρήσης αυτών των μετρητών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ωραία. Κλείνουμε τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ όλους σας. Δίνω και πάλι το λόγο τον Επίτροπο κύριο Γκίντερ Έτιγκερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξάρτητες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω στον κύριο Σβόμποντα ότι η εφαρμογή ε, ο κ. Φόβοντα είπε ότι η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται περιφερειακά. Και πράγματι έχουμε πολύ καλέ εμπειρίε μέχρι στιγμή με προγράμματα εξυγίανση. Πολύ συχνά με ένα ευρώ από δημόσιο προπολογισμό μπορούμε να πετύχουμε ε, πολύ θετικά αποτελέσματα. Ε, μέσω ιδιωτικής επενδυτικής ε, δέσμευσης. Θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο τα περιφερειακά μας ε, προγράμματα μπορούν πράγματι να εφαρμοστούν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει ε, να αξιοποιούνται τα περιφερειακά προγράμματα να ανοίξουν σε σχέδια εξυγίανσης ή ανεκαίνησης των κτηρίων. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο. Ε, όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων, ε, και αυτό είναι σημαντικό, θα πρέπει να υπάρξει μείωση επιτοκίων για δάνεια τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση κτηρίων. Όσον αφορά τα κτηριακά αποθέματα, θα ήθελα να πω ότι ελέγχθη ότι όταν αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση εξοικονομούμε χρήματα. Αυτό ισχύει, αλλά όχι άμεσα. Εάν δούμε την ευημερία στην Ευρώπη, ε, κατά μέσο όρο ανακατοικία έχουμε μια ανάγκη εξυγένσης ή ανακαίνησης από τα παράθυρα μέχρι ε, διάφορες ηλεκτρικές συσκευές ή μέχρι διάφορα θερμαντικά σώματα και την βελτιστοποίηση 30 έως 60.000 ευρώ χρειαζόμαστε ανακατοικία. Και αυτό το, αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα εξοικονομήσουμε τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να επενδύσουμε τα επόμενα 10 χρόνια, ούτω ώστε τα επόμενα 40 χρόνια να μειωθούν οι δαπάνε ε, για την ενέργεια και να υπάρξει επανεπένδυση. Η δική μου γενιά μέχρι τώρα έκανε χρέη για πρώτη φορά έχουμε τώρα την ευκαιρία εμείς να επενδύσουμε στην ενεργειακή απόδοση, ούτω ώστε εμείς και τα παιδιά μας τις προσεχείς δεκαετίες να δουν τα κέρδη μέσω ακριβώς μείωση των δαπανών στην ενέργεια. Είμαστε σε θέση να το κάνουμε, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε. Εγώ πραγματικά υπολογίζω σε εσά. Θα πρέπει σε θέματα προπολογισμού να θέσουμε νέε προτεραιότητε. Όποιος επιθυμεί μια ενεργειακή εξυγίανση και ε, ως προτεραιότητα του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα πρέπει να επίση να συζητήσει, να διαθέσει να συζητήσει τι θα πάει πιο κάτω ε, που θα πρέπει να γίνει, πώς θα πρέπει να γίνει η αναδιάθεση των προτεραιοτήτων. Το θέμα λοιπόν αυτό θα πρέπει να τεθεί ε, στο επίπεδο της ε, κατάρτισης του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Δεύτερον, δύο συνάδελφοι, ο κ. Ζαμπό και ο κ. Άικχαουτ, είπε ότι οι κατευθυντήριες, οι βασικές γραμμές είναι ξεκάθαρες. Όχι, δεν είναι ξεκάθαρες. Και εγώ έχω το, ε, τις αποφάσεις, την τελευταία απόφαση του Συμβουλίου το Μάρτιο αυτού του έτους, επιλέξει και κινούμενοι προς μια αύξηση της τάξης του 20% στην ενεργειακή απόδοση. λέει ότι πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση του 20%, δηλαδή και το 19% και το 18% και το 14% είναι εντάξει. Εγώ θεωρώ το 20% έχει αποφασιστεί και οτιδήποτε άλλο κάτω από αυτό συνιστά οπισθοχώρηση. Ε, το Μάρτιο του 2007 η απόφαση λέει για α, ε, μια προβολή στο μέλλον προοπτική της α, ε, δαπάνης και μια μείωση του 20%. Οι αριθμοί αναφέρονται σε τρεις στήλε. Βλέπετε τι πρόβλημα έχουμε μπροστά μας. Ενεργική κατανάλωση στην Ιταλία σε εκατομμύρια τόνους. Το 2007 173. Το 2020 υπάρχει μια τεράστια αύξηση και θα πρέπει να, να έχουμε μια μείωση του 20%. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση στην ε, ε, προβολή ε, στην πρόγνωση για το μέλλον και μετά βάζουμε το μείον 20%. Στο Λουξεμβούργο επίσης ε, γίνεται αυτή η ε, μελέτη της προοπτικής. Η Πορτογαλία πηγαίνουμε στο 30% και στη συνέχεια κατεβαίνουμε στο 23%. Αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε τι γίνεται για την κάθε χώρα. Ποια είναι, η προοπτική της εξέλιξης και τι γίνεται με τους αριθμούς εάν ε, προσθέσουμε την ε, μείωση του 20%. Εάν θέλουμε να θέσουμε ένα δεσμευτικό στόχο για την κάθε χώρα μέλος, Ε, η πρόταση αυτή θα απορριφθεί σαφώς από τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό προτείνω δύο, ένα πλάνο δύο σταδίων που θεωρώ ότι είναι πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή θα πω στις χώρες μέλη ε, κάντε τα εθνικά σας σχέδια για την ενεργειακή απόδοση, εθελούσια και αν σε δύο χρόνια διαπιστώσετε ότι δεν προχωράτε τότε θα πρέπει να εξαγγείλετε την ε, διατύπωση ε, δεσμευτικών στόχων. Γιατί αυτό δεν θα μπορούν να το απορρίψουν οι χώρες μέλη. Και παρακαλώ να εξετάσετε κατά πόσο αυτό... Ε, κατά πόσο αυτή, αυτός δεν είναι ο ανδεδειγμένος δρόμος και με τη συνένεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την επίτευξη των ευρωπαϊκών μας στόχων. Και όπως είπα, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι στόχοι είναι δεσμευτικοί ή θελούσιοι, τα εθνικά σχέδια δράσης απαιτούνται. Και από πολιτική άποψη μπορούμε να θέτουμε τα περιεχόμενα και τις συνέπειες ή να τα εξετάζουμε τα περιεχόμενα αυτών των σχεδίων, αυτών των πλάνων και τις συνέπειές τους. Ε, και βεβαίως ε, δεν θα αποδεχθούμε κανένα τέτοιο σχέδιο, εθνικό σχέδιο, το οποίο να μην ανταποκρίνεται στους πολιτικούς μας στόχους. Ευχαριστώ πολύ. Όταν παριστώ πάλι στο Κοινοβούλιο θα υποβάλω επισήμως μία πρόταση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τέτοια ώρα που είναι θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή κύριο Μπένστον. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση και όλους τους συναδέλφους που ήταν παρόντες εδώ. Φαντάζομαι ότι ε, καταλάβατε ότι υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις ως προς την ε, δεσμευτικότητα ή όχι, αλλά όχι ως προς το ότι η ενεργειακή απόδοση είναι θετική. Πιστεύουμε ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί, αλλά θα πρέπει να τηρηθούν οι υφιστάμενες ε, νομοθεσίες στην Ένωση. Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για πολλούς νόμους, μετά όμως θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των νόμων. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει κάτι και για τα κτίρια, κάτι για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, για μια καλύτερη πολιτική για τα προϊόντα και για τις μεταφορές. Ε, τελευταία παρατήρηση είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει χρηματοδότηση, κατάλληλη χρηματοδότηση και στο μέλλον. Πολλά πράγματα έχουμε ακόμα να κάνουμε που μπορούμε να πετύχουμε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα, την ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη. Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Κάρινς, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Η Ευρώπη πληρώνει πάμπολα και προς τη Ρωσία και προς τη Μέση Ανατολή. Τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαφώς καλύτερα στην Ευρώπη και είναι σίγουρο ότι αν θέλει η Ευρώπη να είναι ο πρώτος που θα κινηθεί, ο first mover, πρέπει να επενδύσει. Να επενδύσει με μεγαλύ, σε μεγαλύτερες, σε περισσότερες θέσεις σε πιο καινοτόμες επιχειρήσεις, σε καλύτερες δομές ε, λειτουργία των επιχειρήσεων. Επαναλαμβάνω ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στη συζήτηση. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο και τις υπηρεσίες του που έδειξαν εξαιρετική διάθεση συνεργασία και ευχαριστώ και την ομάδα μου που έδειξε την εμπιστοσύνη της σε μένα υποστηρίζοντας τις εργασίες μου για την σχετική έκθεση. Ευχαριστώ er για την εξαιρετική συνεργασία σας. Είναι σημαντικό στη φάση αυτή να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε τόσο ώστε να πετύχουμε ένα πραγματικά ουσιαστικό και ουσιαστικό, ένα πραγματικό και ουσιαστικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Μπένσεν, ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ επίτροπε. Φτά, τελείωσε η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 και περνάμε